Morning, dear colleagues. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό τριμερή διάλογο που λαμβάνει η χώρα και γι' αυτό ήμασταν όλοι εκεί. Σας παρακαλώ να κάνουμε μία δοκιμή για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ο κύριος Καλβέ Σαμπό δεν έχει κάρτα. Τι διαδικαστικό θέλετε εσείς. Όχι. Λοιπόν, δοκιμή είπαμε. Α, ναι, το διαδικαστικό σας. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει καθόλου να παίζουμε ούτε με το χρόνο των βουλευτών, ούτε με τις ψηφοφορίες. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Έχουμε όλοι κάνει μεγάλες προσπάθειες για να είμαστε εδώ στην ώρα μας. Άλλοι πρέπει να φύγουν νωρίτερα, γιατί περίμεναν ότι θα έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Είμαστε πολλοί εδώ για να αρχίζουμε στην ώρα μας και εσείς δεν κάνατε τα απαραίτητα για να ψηφίσουμε σήμερα στην ώρα μας. Δεν είναι δημοκρατική αυτή η διαδικασία, γι' αυτό εγώ προτείνω να μην ψηφίσουμε. Τώρα να ψηφίσουμε μια άλλη μέρα. Πρόεδρος, ζητώ πραγματικά συγγνώμη γιατί βλέπετε παράλληλα είχαμε άλλε συναντήσεις, τον τριμερή διάλογο και δεν θα ήταν οι άλλοι συνάδελφοι εκεί, δεν μπορούσα. Τώρα είμαστε εδώ πέρα, εδώ και συνάδελφοι, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Και αρχίζουμε με την πρώτη ψηφοφορία που είναι η προσωρινή συμφωνία σχετικά με τις υποχρεώσεις OTC, η έκθεση του κύριου Λάγκεν. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. 36 υπέρ, ένας κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Δεύτερη ψηφοφορία. Κριτήρια έκθεση Νίνα Γκίλ. Ψηφίζουμε μονομαστική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 38 υπέρ, κανείς κατά μία αποχή. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Επόμενο θέμα. Συμφωνία για εποπτεία και τα λοιπά για ειδικού φόρους. Ψηφίζουμε, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 39 υπέρ, ομόφωνα. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Επόμενο θέμα. Αποτελέσματα τριμεριού διαλόγου για τις μικρομεσές. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. 36 υπέρ, κανείς κατά, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. Τώρα πάμε στην ψηφοφορία Φερνάντες για τα ESBs. Πρόταση για απόρριψη πρώτα απ' όλα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η απόρριψη. Οπότε συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική Α. Α, 19 ήταν κατά και 12 υπέρ και 8 αποχές είχαμε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οπότε υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική CAA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική CA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική DD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DF e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική DI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και Υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική όχι, πρώτα η 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική R, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική S, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική T, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική U, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική V, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική W, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική WA, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική X, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της τροποποιημένης πρότασης με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 12 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα εδώ και ευχαριστώ και όλες τις πολιτικές ομάδες για την επικοδομητική του στάση. Τώρα, τελειώσαμε. For Τελειώσαμε πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια παράπονα, αλλά όχι πολλά. Announcement for George. Λοιπόν. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις ε, για τις αποφάσεις ε, των συντονιστών. Brexit, έχουμε την ε, διαδικασία μία αντίρρηση τίποτα συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Ο ορισμός αποφασίστηκε τρία θέματα φορολογίας δεν θα δοθούν πριν από το τέλος της θητεία. Ο πρόεδρος έθεσε το θέμα του σπασίματος της πρότασης για τα κόκκινα δάνεια μετά την ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκε ότι θα παρουσιαστούν γραπτός όλες οι επιλογές. Συνεδρίαση των Επιτροπών Ιούλιο Δεκέμβριο εγκρίθηκαν αντιπροσωπείε και επισκέψεις Δουβλίνο Bundesbank. και σύνθεση των επιτροπών ε, το θέμα του Δημοσιονομικού Συμφώνου αποφασίστηκε ότι θυμά αυτά είναι η προηγούμενη συνεδρίαση ομάδα εργασίας ε, χρηματοπιστωτικής βοήθειας συμφωνήθηκε να έχουμε δύο συνεδριάσεις πριν το τέλος τη συνάντηση με τον Ασόκα Μόντι, παρουσία σε τεχνικές επιτροπές, ε, είτε ένας βοηθός είτε ένας σύμβουλος από κάθε ομάδα θα μπορεί να πάει σε ομάδες ε, φυσκάλης, καλυμμένα ομόλογα και benchmarks, Συντονιστέ 26 Φεβρουαρίου η εισηγητή ε, τη ΕΚΟΝ για τον προβλησμό 2020 ΕΛΚ ε, και το προ την προτινόμενη μορφή για τη συνάντηση με τον κύριο Μόντιν και τη Κομισιόν εγκρίθηκε. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόγραμμα εργασίας 2020. Η μεγάλη πλαισία των συντονιστών ενέκριναν το θέμα που πρότεινε ο συντονιστής του ΕΛΚ. Οι τρεις δηλαδή εποπτικές αρχές θα έχουν κάποιες δαπάνες σχετιζόμενες με το Brexit, οπότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά αυτές τις δαπάνες, διαδικασία επίσημων γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Γραμματεία σε διαβούλευση με τον συντονιστή του ΕΛΚ θα προετοιμάσει ένα σχέδιο σύσταση για την επόμενη Επιτροπή με γραπτή διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποια συνέχεια για το ψήφισμα Β80589 του 2018 Τώρα εξέταση πράξεων κατεξιοδότηση από τις 21 Μαρτίου μετακινήθηκε στις 2 Απριλίου και για την προσέλευση στις τεχνικές συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος σοσιαλδημοκρατών συμφωνήθηκε ότι είτε ένας βοηθός είτε ένας σύμβουλος ομάδα θα μπορούσε να πηγαίνει στις τεχνικές συναντήσεις. Αυτά. Τώρα περνάμε στις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις ΕΜΙΡ 2.2 και δηλώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας. Όπως ξέρετε από χτες είχαμε διαλόγους για τον ΕΜΙΡ 2.2 και καταλήξαμε σε προσωρινές ε, συμφωνίες. Ειδικά το Κοινοβούλιο θα επέλεγε υποψηφίους για ανεξάρτητα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής της ε, ΕΣΜΑ η συμφωνία για το άρθρο 22 της ε, ΕΚΤ ε, υπάρχει αλλά έχει ξεπεραστεί από την απόφαση της ΕΚΤ να αποσυρθεί η ΕΣΜΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο Οπότε το πεδίο εφαρμογή πλέον περιορίζεται μόνο σε τρίτες χώρες και άλλα στοιχεία. Πρέπει να πω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είχε ε, καταλήξει αυτή τη σύγκρουση με την ΕΚΤ. Οπότε υπάρχει και μία δήλωση σήμερα σε ένα άρθρο στο Financial Times ε, Δεν ικανοποιηθήκαμε από τη σκληρή στάση του Συμβουλίου και η Κομισιόν δεν έπαιξε επίσης ε, κάποιον εξορροπητικό ρόλο. Τώρα, μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, και η ανάπτυξη, οι αναπτυσσόμενε αγορέ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τις κύριες πρωτοβουλίες, προτεραιότητες του Κοινοβουλίου όπως παραδείγματος χωρίς να καλυφθούν όλες οι επενδύσεις, όχι μόνο αυτές οι οποίες θεωρούνται εφόρο. Τώρα για το ESFS και την εξέτασή του έχουν γίνει πολύ τριμερείς διάλογοι και είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και, και ακριβώς βρισκόμασταν πριν από λίγα λεπτά και θα επαναλάβουμε τις τελικές διαπραγματεύσεις μετά την συνεδρίαση της ΕΚΟΝΕΝΕ. Ναι, ναι. Τέλος, χτες καταλήξαμε σε προσωρινή συμφωνία για το Invest EU και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, τον συνεισηγητή και τους συναδέλφου ε, του προϋπολογισμού για τη στενή συνεργασία. Καταλήξαμε σε μια καλή συμφωνία. Περιλάβαμε πολλές από τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Οπότε, εργαζόμαστε πολύ, όπως βλέπετε και καταλήξαμε σε όλα τα θέματα στα οποία μπορούσαμε να καταλήξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και το προσωπικό για τη δουλειά που έχουν κάνει. Οπότε, μετά, έγκριση των πρακτικών 26-27 Νοεμβρίου, 6 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 21-22 Ιανουαρίου, 21 Φεβρουαρίου, 4 Μαρτίου, 11 Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Και τώρα... ξεκινάμε εγκαίρως την πρώτη δημόσια ακρόαση μετά από την εκλογή του ως επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου με τον Ανδρέα Ενρία. Καλώς ήρθατε. Thank you to, uh, Andrea ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε. Χαιρόμαστε και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας με τον κατάλληλο αριθμό δηλώσεων και για την διαφάνεια πράγματα τα οποία έχετε ανακοινώσει στο Κοινοβούλιο και τώρα ξεκινάει ο καθορισμός αυτής της ε, προσέγγισης οπότε χωρίς ε, περαιτέρω έχετε τον λόγο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ε, πολύ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία σήμερα να σα μιλήσω εδώ πέρα και να σα παρουσιάσω την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, για το 2018. Καθότι είναι η πρώτη μου επίσημη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τελευταία φορά για τη θητεία αυτή, θα ξεκινήσω από κάποιε προσωπικέ εντυπώσει. Κατόπιν θα επικεντρωθώ ε, στα όσα έχουμε μάθει από την δημιουργία τη τραπεζική Τραπεζικής Ένωσης πριν πέντε χρόνια. Θα αναφερθώ σε δύο κυρίως ε, τομεί: ε, το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων και την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων στην ε, Τραπεζική Ένωση. Και θα κλείσω με παρατηρήσεις για τις εποπτικές μας προτεραιότητες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για το 2019, καθώς και την προετοιμασία του Brexit. Ξεκινώντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα και την αφοσίωση του προσωπικού μεγάλος όγκος ε, εργασίας ε, διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα σφιχτά ε, χρονοδιαγράμματα και λαμβάνοντας υπόψη το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που σε πολλούς τομείς απαιτεί ακόμη την εφαρμογή εθνικών κανόνων. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα όταν έρχεται απ' έξω. Ούτε εγώ μπορούσα που είχα πολύ πείρα όσον αφορά την εποπτεία ευρωπαϊκών τραπεζών ξεκινώντας από την ε, αρχική φάση σε μια πιο όρημη φάση, θα απαιτήσει περισσότερο ε, συντονισμό ανάμεσα στις ε, εθνικές αρχές και το κέντρο, αλλά θα οικοδομήσουμε πάνω σε μια πολύ στιβαρή βάση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τότε που δημιουργήθηκε η Τραπεζική Εποπτεία το 2014 έχουμε προοδεύσει σημαντικά όσον αφορά την ποιότητα και την ε, συνεκτικότητα της ε, Τραπεζικής Εποπτείας στον τομέα του ευρώ. Για παράδειγμα, έχουμε ε, εισάγει μια διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγηση σε που μας επιτρέπει την συνεπή αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και έχουμε εναρμονίσει την εφαρμογή 130 ε, επιλογών ε, και που είχαν οι εθνικές αρχές. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει ένα ε, φιλόδοξο έργο, την στοχευμένη αναθεώρηση των εισιτορικών μοντέλων. Αυτή η στοχευμένη αναθεώρηση έχει βοηθήσει στην κοινή κατανόηση των ε, νομοθετικών απαιτήσεων και επιπλέον ε, μας έχει επιτρέψει να διαπιστώσουμε ποια είναι τα ελαττώματα των εσωτερικών μοντέλων που χρησιμοποιούν ε, διάφορα, διάφοροι σημαντικοί φορείς. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο εποπτικό πλαίσιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αποτελείται από τρία στοιχεία. Καθοδήγηση προς τις τράπεζες, όπου έχουμε ε, τις ε, προσδοκίες ως προς την ποιότητα των ε, δανείων, ένα πλαίσιο για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αποτελείται από δύο σκέλη. Πρώτον, αξιολόγηση των στρατηγικών των τραπεζών και σωστή εποπτεία. Και τέλος, ε, ένα παράρτημα στην καθοδήγηση όσον αφορά τα δάνεια αυτά, όπου αναφέρονται ποσοτικές προσδοκίες εποπτείας. Και πράγματι ο όγκο των δανείων αυτών ε, στους ισολογισμούς των τραπεζών ε, έχει μειωθεί από ένα τρισεκατομμύριο αρχέ του 2015 σε 628 δισεκατομμύρια στο τρίτο τρίμηνο του 2018. Παρόλα αυτά είναι υψηλό ο συνολικός όγκος των δανείων ε, αυτών και συνεχίζεται να αυξάνεται και το ποσοστό τους κυμαίνεται μάλλον το ποσοστό τους. Οι δράσεις μας ε, λοιπόν στόχο έχουν να κάνουν πιο ανθεκτικό τον τραπεζικό τομέα. Τα ποσοστά ε, κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ε, έχει αυξηθεί από 11,3 τέλη του 2014 στο 14,1 το 2018. Έχει γίνει πιο σταθερή και η χρηματοδότηση και η ρευστότητα και ενώ έχουν επιτευχθεί πολλά ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμη δεν έχουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς ε, μια ενιαία ολοκληρωμένη ενωμένη αγορά που θα είναι προστατευμένη από ιδιάζουσες κρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε περισσότερο σε κανονισμούς παρά σε οδηγίες και να μειώσουμε τα νομοθετικά ε, εμπόδια στην ε, διασυνοριακή τραπεζική δραστηριότητα όπου αυτό είναι δυνατόν. Ε, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης. Η δημιουργία μιας Τραπεζική Ένωση που λειτουργεί σωστά σημαίνει όχι μόνο μείωση της πιθανότητα μιας τραπεζικής κρίσης, σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αυξήσουμε το δυναμικό αντιμετώπισης των κρίσεων όταν ε, υπάρξουν. Και ε, η τραπεζική εποπτεία έχει δημιουργήσει ε, ένα πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων το οποίο μας ε, επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά ε, τέτοιες καταστάσεις. Το πλαίσιο καθορίζει μια σωστή διαδικασία, μια σωστά καθορισμένη διαδικασία που αποτελείται από διάφορα στάδια. Σε κάθε στάδιο αναλαμβάνονται συγκεκριμένε δράσεις ε, κατάλληλες για την κατάσταση και ιδιαίτερα παρακολουθούμε τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της τακτικής αξιολόγησής τους. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι η τραπεζική εποπτεία καθώς και το Συμβούλιο Ενιαίας, ε, ε, ε, Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης έχουν συνάψει συνεργάζονται στενά σε καθημερινή βάση και επίσης ε, έχει αναθεωρηθεί το μνημόνιο κατανόησης που ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2018. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο. Από νομοθετικής πλευράς απαιτούνται βελτιώσεις ε, για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των μέτρων. Και η επικάλυψη μεταξύ των μέτρων εποπτείας και των μέτρων έγκαιρης ε, παρέμβασης θα πρέπει να εξαλειφθούν. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει νομική βάση κανονισμού για τις ε, εξουσίες ε, έγκαιρης παρέμβασης ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων μάλιστα δημιουργήθηκε για να καλύψει κάποια από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Περνάω τώρα στην νομοποίηση παράνομων εσόδων. Ένα πράγμα μάθαμε από την ε, χρηματοοικονομική εποπτεία το 2018, ότι απαιτείται περισσότερη βελτίωση στον τομέα της καταπολέμησης νομοποίησης παράνομων εσόδων. Παρότι ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι αρχή με αρμοδιότητα την ε, καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων, βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα για τον τομέα αυτό και εσύ πρόσφατα ε, συνάψαμε συμφωνία με τους ε, εθνικούς επόπτες ε, στον ΕΟΧ που είναι αρμόδιοι για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Επιπλέον, ο προκάτοχός μου πέρσι ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσουμε μία λειτουργία συντονισμού στον ε, τομέα αυτό και θα συντονίζουμε τις εργασίες ε, των ε, κοινών εποπτικών ομάδων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα αυτών και γι' αυτό χρειάζεται η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να ενισχυθεί το πλαίσιο για το, την καταπολέμηση των προβλημάτων στον τομέα αυτό. Κατόπιν, ε, θα ήθελα να σα ενημερώσω σχετικά με τις εποπτικές ε, προτεραιότητε μας για το 2019. Καταρχά, θέλουμε μείωση του όγκου των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, ως μέρος μιας νέας πρωτοβουλία θα εξετάσουμε τις, τα ανοίγματα των τραπεζών και έτσι θα εξετάσουμε την ε, ποιότητα των ε, ανοιγμάτων των τραπεζών. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, διαχείριση κινδύνου, θα, θα συνεχίσει το TRIM που σας ανέφερα, που είναι η στοχοθετημένη αναθεώρηση εσωτερικών μοντέλων. Θα εξετάσουμε επίσης και θα συνεχίσουμε να προωθούμε βελτίωση στις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών όσον αφορά την κεφαιρειακή επάρκεια και την επάρκεια σε ρευστότητα. Τέλος, οι εποπτικέ δραστηριότητε για το 2019 συμπεριλαμβάνουν εργασίε που έχουν να κάνουν με του κινδύνου. Ε, στο εμπόριο και την ε, αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώ και προετοιμασία του Brexit που θα συζητήσω τώρα. Το Brexit ε, ήταν προτεραιότητα για μα τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά την εποπτεία και υπάρχει σημαντική βεβαιότητα όσον αφορά τα επόμενα βήματα στην διαδικασία αυτή. Η παρούσα στιγμή φαίνεται να μην έχει αποκλειστεί η λύση του σκληρού Brexit και έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για να προετοιμαστούμε και έχουμε πιέσει και τις τράπεζες να προετοιμαστούν για κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Έχουμε αξιολογήσει διάφορες αιτήσει ε, αδειών από τράπεζες που θέλανε να, με, μετικήσουν στην περιοχή του ευρώ και έχουμε δώσει άδεια σε όλες τις τράπεζες που ε, ε, υπέβαλαν αίτηση εγκαίρως. Επίσης, έχουμε συνεργαστεί στενά με διάφορους ετούντες για να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μέτρων επίγουσας κατάστασης. Επιπλέον έχουμε εξετάσει τα σχέδια των ε, τραπεζών ε, που έχουν έδρα εντός ε, της ζώνης του ευρώ. Ανάλογα με τον βαθμό που εξαρτώνται από τις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να υπάρξουν κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την μετάβαση σε ένα περιβάλλον με Brexit. Όσον αφορά την ε, εποπτική μας ε, στρατηγική, συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα ε, στιβαρό πλαίσιο για τη συνεργασία μετά το Brexit. Και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει συντονίσει με επιτυχία ένα σχέδιο για την συνεργασία αυτή. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το PRA από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συμφωνήσει όσον αφορά τον διαχωρισμό των ε, αρμοδιοτήτων εποπτείας, όσον αφορά τις ε, τα διάφορα καταστήματα, υποκαταστήματα των τραπεζών. Επίσης έχουμε ξεκινήσει εσωτερικές προετοιμασίες ε, για να προετοιμαστούμε για το Brexit και βέβαια παρακολουθούμε στενά και την εφαρμογή από τις τράπεζες των ε, σχεδίων επίγουσας κατάστασης ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε αν υπάρχουν καθυστερήσεις. Και θα κλείσω τα τελευταία πέντε χρόνια τα πρώτα πέντε χρόνια τη ε, τραπεζική εποπτεία ε, στην Ευρώπη. Έχει δημιουργήσει συνθήκε ίσου ανταγωνισμού για τι ε, τράπεζε στη ζώνη του ευρώ και έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα του τομέα. Απομένουν όμω πολλά να γίνουν ακόμα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τα όσα μάθαμε από την κρίση, ούτε θα πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό να χαλαρώσουμε του κανόνε μόλι βελτιωθεί η κατάσταση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ικανό, επικριτικό και χρήσιμο εταίρο για την τραπεζική εποπτεία κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία σε Προσλέπω στην ε, συνέχεια της συνεργασίας ε, μαζί σας μετά τις επικείμενες ευρωεκλογέ. Και πολύ ευχαρίστω θα απαντήσω σε ερωτήσεις και θα ακούσω σχόλια. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ανδρέα Ανδρία, για την παρουσίασή σας, για όλα τα θέματα που θίξατε. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις για σας, αλλά ο Μάρκους Φέρμπερ είναι ο πρώτος που έχει ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ενρία. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ με τη νέα σας ιδιότητα. Ε, αν και θα χαιρόμουν να, δω και γυναίκα στη θέση σας, αλλά φυσικά τελικά αποφασίζει η πλειοψηφία. Ε, δύο σύντομε ερωτήσει. Αναφερθήκατε στην καταπολέμηση τη νομοποίηση παράνομων εσόδων. Ε, ο προκάτοχός σας είχε ανακοινώσει την δημιουργία γραφείου ε, για την καταπολέμηση του ε, ξεπλήματος χρημάτων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι ακριβώς γίνεται στον τομέα αυτόν. Επίσης, η προηγούμενη σας αρχή, ο ενιαίος επιτοπτικός μηχανισμός είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό και είχαμε και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, τραπεζών όπως είναι η ABN. Θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις σας για το θέμα αυτό. Δεύτερον, ε, όσον αφορά το μεγάλο ποσοστό ε, δανείων κρατών στο στο χαρτοφυλάκιο διαφόρων τραπεζών. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρέπει, συγγνώμη, για, το, για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Πρέπει να σας πω ότι ναι, η λειτουργία αυτή έχει εγκριθεί στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι προσλαμβάνουμε προσωπικό, άρα θα αρχίσει τις λειτουργίες του το σώμα αυτό πολύ σύντομα. Αλλά θέλω και να διευκρινίσω ποιος είναι ο ρόλος που έχουμε εμείς, ο εποπτικός γιατί φυσικά και αυτά τα θέματα τα περιλαμβάνουμε στους ελέγχους μας. Αλλά όπως είπα και στις αγωγικές μου παρατηρήσεις, υπάρχουν διαφορετικοί τομείς όπου μπορεί να είναι χρήσιμη η δικιά μας η δουλειά. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε ζητήματα ε, στη δικιά μας την εποπτεία, τη συνήθη της ρουτίνας και έχουμε ένα πλαίσιο και έχουμε και ε, συμφωνία με τις ε, εθνικές αρμόδιες αρχές προκειμένου ότι οι πληροφορίες υπάρχουν να φτάνουν ε, στους αρμόδιους επόπτες κατά της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Τώρα είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις άδειες της τράπεζες και κάνουμε αξιολόγηση εκεί που πρέπει και είμαστε αυστηροί όπου πρέπει να είμαστε αυστηροί ώστε να μην εισέρχονται στο σύστημα των ευρωπαϊκών ε, τραπεζών τέτοιοι κίνδυνοι. Υπάρχει διακυβέρνηση, υπάρχει εσωτερικός έλεγχος. Κάθε τράπεζα η οποία έχει σοβαρά προβλήματα με το ξέπλυμα χρήματος ή που δείχνει αδυναμίες στην διακυβέρνηση και στους εταίρους ελέγχους εντοπίζεται αμέσως από εμά. Οπότε ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τις αρχές καταπολέμησης παράνομων ε, εσόδων. Βοηθάμε εμείς αυτούς και εκείνοι εμάς. Και από την άλλη ενισχύουμε και την ε, προσοχή μας σε αυτά τα θέματα όταν προβαίνουμε στους τακτικούς μας ε, μακροπροληπτικούς ελέγχους. Τώρα, για το θέμα της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Τραπεζών στα, στο δημόσιο χρέος. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν υπάρξει ανησυχίες στο παρελθόν και όντω υπήρξαν τράπεζες οι οποίες ήταν υπερβολικά εκτεθειμένες. Ε, θυμάμαι ότι είχα δει τα ποσά και μερικές φορές είχαν πάνω από 10% από το επιτρεπόμενο. Και αν αυτά τα μέσα, αυτοί οι μηχανισμοί ήταν ε, όπως έπρεπε, φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούν το κεφάλαιο που διαθέτουν σαν ε, ε, μέσο προστασίας σε περίπτωση κρίσης για τη ρευστότητά τους. Οπότε η υπερβολική συγκέντρωση πράγματι είναι ένα ζήτημα και θα έπρεπε να το κοιτούμε κι εμείς κάθε φορά που προβαίνουμε σε ελέγχους. Ωραία, πολύ ωραία τα λέτε, αλλά πιο συγκεκριμένα Μα είναι σαφές ότι αν ε, βλέπετε ότι υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση, τότε ζητάτε από την τράπεζα να το αλλάξει, να το φροντίσει. Και στο παρελθόν, θυμόσαστε ότι μία από τις πρώτες δράσεις μου το 2011, όταν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και υπήρχε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκών τραπεζών υπερβολικής έκθεσης στο δημόσιο χρέος, ε, τους ζητήσαμε να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Και ζητήσαμε να υπάρξει στον πυλώνα 2 ένα σύστημα κεφαλιακής προστασίας για να μην ε, επαναληφθεί το φαινόμενο ξανά. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Θα επικεντρωθώ εγώ σε τρία ζητήματα. Πρώτον, μας υπενθυμίσατε το πλαίσιο για τα NPL για το νέο πλαίσιο, για αποθέματα και κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις, μάλλον μία ερώτηση. Όσον αφορά το απόθεμο, σωστά λέτε ότι αποτελεί μέρος του παπτικού διαλόγου και των προσδοκιών των τραπεζών. Οπότε πράγματι αυτό που αποφασίστηκε τον Ιούλιο ήταν να υπάρχει διάλογος ε, δηλαδή δράση και αντίδραση και οι εποπτικές ε, προσδοκίες θα είναι πολύ συγκεκριμένες για τις τράπεζες. Από αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό το επιβεβαιώνεται. Δεύτερον, κάτι πιο δύσκολο, γιατί τώρα έχουμε ολοκληρώσει διαπραγματεύσει για τον πρώτο πυλώνα, για τον, ε, την προληπτική προστασία αλλά τώρα υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στις ε, προσδοκίες της εποπτείας και του πυλώνα αυτού. Και μπορεί να υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον πρώτο πυλώνα και το δεύτερο πυλώνα, αλλά άλλο είναι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εξατομικευμένες και άλλο είναι γενικά να υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες κανόνων από την εποπτική αρχή. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Και ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου χτες που όπως πάντα ζητούσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι οι εγγύησει καταθέσεων πρέπει να προβλεφθούν και για προληπτικούς λόγους βάσει του 11.3 της ανάλογης οδηγίας. Και ήταν κάτι που το έχουμε πει και εμείς ξανά και ξανά. Γιατί Αλλιώς η βοήθεια που δίνεται θεωρείται κρατική ενίσχυση. Όπως ξέρετε οι συνέπειες είναι τεράστιες. Και είναι πολύ επίμαχο αυτό το ζήτημα. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Κούπμαν, ο οποίος είπε, που ήμουν με τον κύριο Σίμων, που είπε ότι η Επιτροπή λέει μα το δικαστήριο Μα αναγκάζει. Αλλά δεν ήταν έτσι, γιατί να, τώρα το δικαστήριο αποφάσισε κάτι εντελώ διαφορετικό. Οπότε εσεί, πώ ε, βλέπετε, τι δουλειά χρειάζεται για να βελτιωθεί το κοινό μα πλαίσιο εξυγίανση. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το πλαίσιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να επιβεβαιώσω την ερμηνεία σας για την κατεύθυνση που δώσαμε για τα ιστορικά αυτά στοιχεία ενεργητικού. Αυτό είναι τμήμα του, του εποπτικού διαλόγου. Αποστέλαμε δηλαδή επιστολές στις τράπεζες και καθορίσαμε κάποιο χρονικό πλαίσιο. Ξεκινήσει τώρα ο διάλογος και θα ενσωματωθεί ε, στην ε, διαδικασία αυτή φέτος και θα Βεβαίω εντός του διαλόγου αυτού οι τράπεζες ε, μπορούν να αμφισβητήσουν την καταλληλότητα των συστάσεων σε σχέση με συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και θα υπάρξει μια συζήτηση και έτσι θα διηγηθούμε στις τελικές προσδοκίες που μετά θα επικοινωνήσουμε και ελπίζω μετά να εκτελεστούν από τις τράπεζες. Για το παράρτημα να πω πως υπάρχει βεβαίως ένα ζήτημα χρονισμού και διαφορετικής εστίασης ε, γιατί η νομοθεσία που έχουν συντάξει οι συνομοθέτες λέει ότι θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε νόμους που ισχύουν αν δεν κάνω λάθος από τον Ιούνιο τρέχοντος οπότε αυτά είναι... υπάρχουν τμήματα του βιβλίου δανείων που δεν θα επηρεαστούν επίσης να υπενθυμίσω εδώ ότι παρά το ότι το πλαίσιο διαμορφώθηκε με αρκετά λεπτόμερη τρόπο δημιούργησε παρόλα αυτά κάποιες εποπτικές προσδοκίες οπότε υπάρχει το ζήτημα του πώς να διαμορφωθεί η μετάβαση από το ένα μέσο στο άλλο ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε βεβαίως οι απαιτήσει πυλώνα 1 επίπεδου 1 θα παραμείνουν ως ε, μια δικλίδα ασφαλείας ε, πυλώνα 1 βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να ζητήσουν επιπρόσθετες ε, δικλίδες επιπρόσθετα μέτρα πυλώνα 2 αλλά βεβαίως εδώ πέρα δεν υπάρχουν κανόνες που επικαλύπτονται Βεβαίως ε, δεν έχουμε κάνει ακόμα μία ανάλυση βάθο, αλλά χτες εκδώσαμε την εποπτική μας έκθεση και είναι σαφές ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι όσον αφορά την διαχείριση κρίσεων και αυτό το οποίο θα έλεγα εδώ είναι ότι τα μαθήματα αυτών των πρώτων ετών για την εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου έχουν δείξει ότι ειδικά στο θέμα αυτό ρευστοποίησης και παρέμβασης των εργαλείων που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις που δεν είναι ευθύνη του ενιαίου μηχανισμού διάσωσης σε αυτούς τους τομείς υπάρχουν ακόμα διάφορες πρακτικές ε, και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ομοιομορφία οπότε ο δυνητικός ρόλος ε, των ε, αρχών αυτών ε, ε, θα μπορούσε να επιτελέσει κάποια λειτουργία στην περίπτωση στην οποία θα έχουμε τράπεζε που θα βρεθούν σε δυσκολίε. Βεβαίω πρέπει να διαβάσουμε προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά τα οποία είπατε για το παράρτημα. Και διάβασα εδώ πέρα τα όσα αναφέρονται προφανώς εάν το ΕΚΟΦΗΝ αποφασίσει μέτρα πυλώνα 1 νομοθετικά μέτρα δηλαδή αυτή τη στιγμή εφαρμοστούν θα εφαρμόσουμε και, θα προσαρμόσουμε και εμείς τα δικά μας μέτρα και τώρα επόμενος μολτής δεν βλέπω εδώ κάποιον από το ECR ή το άλλο οπότε ο Σβέν Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καλώς ήρθατε με τη νέα σας ιδιότητα και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία μας, όπως είχαμε πολύ καλή συνεργασία και στο παρελθόν. Έχω κάποιες συγκεκριμένες και γρήγορες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, στο παρελθόν ήσασταν υπέρ της ε, διαφάνειας ε, των αποτελεσμάτων του πυλώνα 2 και των τον αλλά και υπέρ της δημοσίευση ε, των αποτελεσμάτων ε, των stress test, όπως έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν και στο νέο σας ρόλο θα διασφαλίσετε εάν η διαφάνεια που υπάρχει στον ενιαίο μηχανισμό είναι είναι στο ύψο των προσδοκιών σα. Κατόπιν ε, διαβάσαμε ότι στην αναφορά των κινδύνων δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις μοχλευμένες χρηματοδοτήσεις παρά το ότι υπήρχε μια έντονη προειδοποίηση του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος ε, και γιατί δεν υπάρχει στοιχατογράφηση των κινδύνων. Ε, τρίτον, ε, όταν μιλήσατε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ευχαριστώ που το αναφέρατε, ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε έτσι ώστε αυτά να ισχύουν ε, όχι μόνο για τις αμέσως υποπτευόμενες τράπεζες αλλά και για τις μικρότερες τράπεζες για τις οποίες έχετε ακόμα ευθύνη να διασφαλίσετε παρόμοια επίπεδα ρυθμιστικών προδιαγραφών. Και τέλος, η έκθεση για την ABLV η οποία κινδυνεύει ε, με χρεοκοπία ε, είναι ακατανόητη θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε μια εκδοχή η οποία θα είναι λιγότερο λογοκριμένη για να γίνετε κατανοητή Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θίξατε διάφορα θέματα όσον αφορά τον πυλώνα 2 ε, και το stress test. Θα χρειαζόμουν αρκετό χρόνο για να σας εξηγήσω τι ακριβώς πιστεύω εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Νομίζω ότι οι απαιτήσει του πυλώνα 2 πρέπει να δημοσιεύονται. Συνδέονται με το μέγιστο διανεμητέο ποσό και μπορούν να ε, οδηγήσουν στην ε, καταβολή τοκομεριδίων είναι πληροφορίες σε βάση που πρέπει να δημοσιεύονται. Η καθοδήγηση του πυλώνα 2 πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δημοσιεύεται. Δημοσιεύουμε αρκετέ πληροφορίες στην Ευρώπη όσον αφορά το stress test, ε, την ε, Μιλάμε για ε, εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, στοιχεία δεδομένων για κάθε τράπεζα, που, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε δημοσιεύουν μόλις 90. Το θέμα είναι λοιπόν πού θέτουμε τον πύχη της εποπτείας στα κεφάλαια ως αποτέλεσμα των stress test. Αυτέ είναι πληροφορίες που αυτή τη στιγμή δεν δημοσιεύουμε ή τουλάχιστον δεν τι δημοσιεύουμε ε, με εναρμονισμένο τρόπο. Διότι δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι τώρα στη ζώνη του ευρώ έχουμε τράπεζες σε κάποια κρατημέλη που δημοσιεύουν τα πάντα, τις απαιτήσει του πυλώνα 2, την καθοδήγηση του πυλώνα 2, καθώς και σχέδια επιστολών που στέλνουμε στις τράπεζες, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν δημοσιεύονται καθόλου πληροφορίες, ούτε καν οι απαιτήσει του πυλώνα 2. Έχουμε λοιπόν ε, όλο το φάσμα διαφόρων συμπεριφορών. Πρέπει να εναρμονίσουμε τον ε, τρόπο δημοσίευσης ε, των πληροφοριών αυτών. Και πιστεύω ότι πρέπει να δημοσιεύονται και οι απαιτήσει και η καθοδήγηση του πυλώνα 2. Αν και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι επίμαχο θέμα. Στον τομέα της εποπτείας ε, δεν συμμερίζονται όλοι τη θέση αυτή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν δύσκολες συζητήσεις. Όσον αφορά το stress test, αυτή τη στιγμή δημοσιεύουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες, αλλά δεν είναι οι πληροφορίες που τελικά ε, εισάγονται στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, στη διαδικασία SREP. Έχουμε τα στοιχεία αυτά τον Ιούλιο και έχουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας ΕΣΤΡΕΠΕ τον Δεκέμβριο. Και ο τρόπος που συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα αυτά στην τελική διαδικασία επικύλουν ανάλογα με την ε, κρίση του επόπτη. Αν σας ενδιαφέρει, ε, πέρσι έκανα, ε, έκανα μια παρουσίαση στην Ρουμανία όπου αναφέρθηκα ακριβώς στο τέλος της διαδικασίας ΣΡΕΠ και την παροχή ε, των ε, σωστών πληροφοριών στην αγορά. Ποια είναι λοιπόν η αξιολόγηση του ΕΠΟΠΤΗ όσον αφορά την κατάσταση της τράπεζας. Νομίζω ότι αυτές είναι οι χρήσιμες ε, και οι απαραίτητες πληροφορίες και αυτό θα πρέπει να γίνει γενικά για όλες τις τράπεζες. Όσον αφορά το leverage finance, την χρηματοδότηση κατόπιν μόχλευσης, Έχουμε εκδώσει κατευθυντήρε γραμμέ το 2017. Τώρα εξετάζουμε την εφαρμογή των ε, ε, <clears throat> οδηγιών αυτών και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεικτή εικόνα. Διάφορες πτυχές έχουν εφαρμοστεί σωστά από τις τράπεζες και η πιο σημαντική προστιθέμενη αξία ήταν η διαπίστωση του επίπεδου τέτοιας ε, χρηματοδότησης καθώς και η σωστή διαχείριση τέτοιων ανοιγμάτων. Άλλε πτυχέ εφαρμόζονται λιγότερο ικανοποιητικά και εξετάζουμε μαζί με τις τράπεζες ε, τις περιπτώσεις αυτές. Ανησυχούμε επίση ε, διότι δεν έχει, δεν έχει αυξηθεί σημαντικά ο, ο όγκος και δεν ε, φτάνουμε τα παγκόσμια επίπεδα. Νομίζω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάμε για 2,3 τρισεκατομμύρια, ενώ σε ευρωπαϊκό μιλάμε για 310 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε όμως αυξημένη εξάρτηση από συναλλαγές υψηλής μόχλευσης. Έχουμε δηλαδή μόχλευση άνω ε, των, ε, των, των 60 φορών του ποσού αυτού και το 50% αυτών ε, βρίσκονται σε δύσκολη θέση και γι' αυτό έχουμε εκπονήσει κάποια κοινά πρότυπα που ε, αποτελούν καθοδήγηση και για λιγότερο σημαντικές ε, τράπεζες. Δεν ξέρω αν έχει ε, εκδοθεί κάτι συγκεκριμένο για το μέγεθος των τραπεζών. Ναι, μπορώ να επανέλθω με τις πληροφορίες αυτές. Και όσον αφορά την ε, απόφαση για τις ε, τράπεζες που είναι πιθανό να χρεοκοπήσουν, καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Και το θέμα είναι γιατί δημοσιεύουμε κάτι ένα χρόνο μετά τη λήψη της απόφασης. Νομίζω ότι πρέπει να κινούμαστε πολύ πιο κοντά χρονικά στην ε, απόφαση. Νομίζω λοιπόν ε, ότι όσον αφορά το ε, ενιαίο συμβούλιο εξυγίανση ε, πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Όσον αφορά όμω ε, τι λογοκριμένε εκδόσει, ε, εξαρτώμαστε από τα νομικά μας τμήματα και πράγματι πολύ συχνά είναι πολύ πιο λογοκριμένε οι δημοσιευμένε αποφάσει σε σχέση με αυτό που θα θέλανε οι επόπτε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις σύντομα. Πρώτα απ' όλα για τις συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ευρώπη και μάλιστα των πολύ μεγάλων, του Big to Fail. Δεν μπορούμε βέβαια να μπούμε στις λεπτομέρειες, αλλά θέλω τη γνώμη σας για τις συγχωνεύσεις που μπορεί να γίνουν ανάμεσα σε τράπεζες που ίσως έχουν διαφορετικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία. Αλλά φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Οπότε γενικά ποια είναι η άποψή σας αν δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος με τράπεζες του big to fail δεν θα γινόντουσαν ακόμα πιο μεγάλες με τις συγχωνεύσεις αυτές. Και αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, δεν αναφερθήκατε στη δράση για την ρευστότητα. Πάντα είχατε αρνηθεί διαφορετική μεταχείριση κατά περίπτωση. Αλλά σε σχέση με την προηγούμενη διαχείριση, εσείς τι θα κάνετε, θα κάνετε περισσότερα. Και έχω και μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να με καθησυχάσετε παρακαλώ. Όσον αφορά τι τις δοκιμές αντοχής τι θα κάνετε στο μέλλον. Γιατί είχε υπάρξει προσφυγή σε ιδιωτικέ επιχειρήσει, υπήρξε θέμα σύγκρουση συμφερόντων με τα δεδομένα από αυτέ τι δοκιμέ. Μπορείτε να μα διαβεβαιώσετε ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ για τι ε, συγχωνεύσεις. Να πω πρώτα απ' όλα ότι ε, ο στόχος της εποπτείας ε, της ΕΚΤ έχει πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα στην περίπτωση συγχωνεύσεων. Δηλαδή αν μας υποβληθεί η συγχώνευση ε, εμείς πρέπει απλά να αξιολογήσουμε την βιωσιμότητα του εγχειρήματο, εάν έχουν δηλαδή ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχέδιο με τη δυνατότητα κερδοφορίας, ε, ισχυρή διοίκηση με δυνατότητες εκτέλεσης και επαρκές επίπεδο κεφαλαίου και ρευστότητες στο τελικό σχήμα. Δηλαδή όλα αυτά καταλήγουν τελικά στο να διασφαλίσουμε ότι η οντότητα η οποία θα προκύψει θα μπορεί να συμμορφωθεί και να συμμορφώνεται διαρκώς με τις εποπτικές απαιτήσεις. Εκεί εστιάζουμε. Όσον αφορά αυτές που είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν δεν νομίζω ότι γενικώ θα πρέπει να έχουμε μια προκατάληψη κατά του μεγέθους. Το θέμα αυτό σχετίζεται με δύο ρήτρε ασφαλείας. Το πρώτο είναι ότι αν μια τράπεζα γίνει πολύ μεγάλη, πολύ διασυνδεδεμένη, πρέπει να ε, εσωτερικοποιήσει τους κινδύνους ε, τους οποίους αποτελεί. Δηλαδή πρέπει να έχει επιπρόσθετη κεφαλιακή επάρκεια στον ισολογισμό για να μειωθεί η πιθανότητα ε, χρεοκοπίας που θα δημιουργήσει ζημιές στον υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικονομία. πολύ σημαντικά και βεβαίω θα έχει επιπτώσει στι υπόλοιπε συστημικέ τράπεζε και το χρηματοπιστικό τομέα. Και βεβαίω, ε, υπάρχουν και αυτά τα οποία αναφέρονται στην οδηγία περί ε, λύσεις ε, των τραπεζών, δηλαδή και το ότι οι τράπεζες ακόμα και αν φτάσουν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος σε περίπτωση κρίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, να υπάρξει κάποια λύση των τραπεζών δηλαδή μια απλή διοικητική ε, και νομική δομή και δυνατότητα απορρόφησης ζημιών για να βγει από την αγορά αν χρειαστεί η τράπεζα ομαλά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε όταν μιλάμε για συγχωνεύσεις. Μια που είμαστε στο θέμα των συγχωνεύσεων, να πω και κάτι το οποίο δεν ε, ρωτήσατε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί συχνά μιλάμε για εγχώριε, διασυνοριακέ συγχωνεύσει και αν πρέπει να ευνοούμε τι μεν ή τι δε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους βιομηχανικής ας πούμε πολιτικής όσον αφορά τις ε, συγχωνεύσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν πλέον εκτήματα στις εγχώριες συγχωνεύσεις γιατί υπάρχει καλύτερη κάλυψη κόστους και δυνατότητα ε, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας αλλά ε, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις, σε ένα περιβάλλον ρυθμιστικό το οποίο θα ε, ευνοεί δομικά τις εγχώριες ε, συγχωνεύσεις, το οποίο δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα πλαίσιο το οποίο δεν δημιουργεί θετικό περιβάλλον για διασυνοριακέ συγχωνεύσει. Όσον αφορά τα στοιχεία επίπεδου 2, επίπεδου 3, με συγχωρείτε αν δεν ήμουν σαφή στην αρχική μου δήλωση. Πράγματι στι προτεραιότητε του 2019 υπάρχει μια συγκεκριμένη προτεραιότητα για τον κίνδυνο της αγοράς και την αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού που αφορώ ακριβώς το πώς θα πηγαίνουμε πιο πολύ στην ε, ε λεπτομέρεια της αξιολόγησης περίπλοκων στοιχείων του ενεργητικού. Ήδη από την ΕΚΤ είχαμε κάνει κάποιες ε, βαθιές και επιτόπιες αναλύσεις ειδικά σε τράπεζες που ήταν ιδιαίτερως εκτεθειμένες σε αυτά τα περίπλοκα μέσα. Επίσης να αναφέρω για λόγους ε, σαφήνειας πως ε, τα στοιχεία επίπεδου 2 και επίπεδου 3 είναι μια δέσμη πολύ διαφορετικών τέτοιων στοιχείων ενεργητικού, πολύ περίπλοκα, πολύ ε, επικίνδυνα που μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες ε, ρυθμιστικές ανησυχίες και υπάρχουν και κάποια πιο απλά προϊόντα τα οποία παρέχουν οι τράπεζες ε, στους εταιρικούς πελάτες τους και τους βοηθούν σε τέτοιες ε, συναλλαγές. Όσον αφορά τους ε, συμβούλους, πράγματι είμαστε ήδη στο φετινό προϋπολογισμό προβλέπουμε σημαντική αύξηση του προσωπικού μας. Δεν θυμάμαι τους αριθμούς. Νομίζω ότι μιλάμε για 40, 40 άτομα επιπλέον που προσλαμβάνουμε φέτος ακριβώς ε, για να ε, κάνουμε εσωτερική αυτή τη λειτουργία που αφορά τα stress test και να μειώσουμε και ή δυνατόν να εξαλείψουμε ε, την εξάρτησή μας από εξωτερικούς συμβούλους. Σας ευχαριστώ, Ντανούτα Χούπνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη ερώτηση έχω διότι νομίζω ότι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που δώσατε, νομίζω στην Financial Times, όταν σας ρώτησαν σχετικά με τις ανησυχίες σας, αναφερθήκατε ε, στα... Στα, στα δημόσια χρέη μπορείτε να δεχτείτε στον τομέα αυτών ποσοστά συγκέντρωσης ε, ή ε, δάνεια μηδενικού κινδύνου. Τι λύση μπορείτε να προτείνετε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, το έχω σκεφτεί πολύ το θέμα αυτό, διότι όπως ανέφερα πριν, η συγκέντρωση δημοσίου χρέους ε, είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει και μάλιστα ήταν πολύ σοβαρό κάποια στιγμή. Η πείρα μου μου λέει ότι καταρχάς θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή ε, στην λογιστική αντιμετώπιση αυτών των ανοιγμάτων. Μερικές φορές βλέπουμε οι τράπεζες να μεταφέρουν τα ανοίγματα από ε, τους ε, λογαριασμούς τους ε, στο Help to Collect που ε, αναφέρονται τα μέσα με ιστορική αξία και όταν επιδεινώνονται οι συνθήκες ε, στην αγορά και από εποπτικής πλευράς δεν είναι αυτή η θετική εξέλιξη. Θέλουμε τουλάχιστον τα στοιχεία του ενεργητικού που καλύπτονται ε, στο ποσοστό κάλυψης 1,1 ε, ή 1,2 φορές το, το ποσοστό των ε, ανοιγμάτων ε, και όταν δούμε αύξηση του κινδύνου στην αγορά, να έχουμε άμεση κάλυψη από την αγορά. Πάντα ήμουν κατά του ορίου μεγάλων ανοιγμάτων, διότι νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι επιζήμιο. Κάποια κίνητρα όμως κατά της ε, υψηλής συγκέντρωσης ε, θα ήταν επιθυμητό. Και να υπάρχουν και κάποια τέλη όταν το ποσοστό αυτό γίνεται υπερβολικά μεγάλο. Απογοητεύτηκα που στο Συμβούλιο η ιδέα των ασφαλών ευρωπαϊκών ομολόγων, ε, τα καλάθια αυτά εξασφαλισμένων μέσων, δεν έγιναν αποδεκτά. Δεν βρήκανε μεγάλη υποστήριξη. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε όμως, ώστε οι τράπεζες να έχουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό εργαλείο στα χέρια τους που να θεωρείται εξασφαλισμένο στοιχείο του ενεργητικού. Ευχαριστώ, Βίντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ενρία, θα θέσω στα γερμανικά την ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Είπατε ότι κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία έχουν επιτευχθεί πολλά όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και την εξασφάλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπατε όμως ότι χρειαζόμαστε περισσότερα, πρέπει να βασιστούν περισσότερο σε κανονισμούς ε, αντί για οδηγίες. Ε, και ε, σας ρωτώ λοιπόν, σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε άμεσο ευρωπαϊκό δίκαιο αντί για οδηγίες που πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο των κρατών χωρών. Πού θα περιμένατε κάτι τέτοιο και βέβαια δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει το επόμενο κοινοβούλιο. Και επίσης ε, στο Συμβούλιο, στο ΕΚΟΦΗΝ βλέπω να υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο όσον αφορά την ε, εμβάθυνση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και περνώ στο θέμα των εθνικών απόψεων. Έχει αναφερθεί το θέμα αυτό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε. Πώς βλέπετε εσείς την επιθυμία να βασιστούμε στους National Champions. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα γερμανικά μου φαντάζομαι θα βελτιωθούν τώρα στη Φραγκφούρτη, αλλά προς το παρόν. Λοιπόν, Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Σίγουρα υπάρχουν τομείς όπως ε, η κατάλληλη αξιολόγηση που εγώ έχω υπογραμμίσει και υπάρχει δυσκολία να πετύχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πρακτική. Βλέπετε οι πρόεδροι συμβουλίων, ε, τα στελέχη κλπ μένουν στις θέσεις τους. Οπότε έγινε μια προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές, εναρμονισμένες πρακτικές δηλαδή. Αλλά πολλές εθνικές αρχές αισθάνθηκαν ότι δεν ήταν σε θέση να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί πρέπει να εφαρμόσουν εθνική νομοθεσία που τους πήγαινε προς άλλη κατεύθυνση. Εμείς όταν μιλούσαμε για εξάντε ή εξπόστ αξιολόγηση, αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί, το οποίο όμως το εφαρμόσουν πολύ διαφορετικά οι διάφορες χώρες. Και εμείς στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συγκεράσουμε πολλές και διαφορετικές πρακτικές και νομοθεσίες. Οπότε μερικές φορέ αναγκαζόμαστε να πούμε όχι. Αυτό είναι ένα. Το άλλο που είπα και στην αρχή είναι το θέμα των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. Υπάρχει βέβαια κάποια επικάλυψη ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα και τα μέτρα τα προληπτικά εποπτείας που υπάρχουν στον κανονισμό και οι επόπτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από ότι η έγκαιρη ε, παρέμβαση. Οπότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν καλό να είχαμε ένα πλαίσιο πιο έτσι, κατάλληλο και ισχυρό για την έγκαιρη παρέμβαση. Τώρα το άλλο. Υπάρχουν διαφορές στις χώρες μέλη. Ας πούμε υπάρχει ο δανέζικος συμβιβασμός στο πρώτο κύμα. Κάτι το οποίο άφησε μεγάλα περιθώρια διακριτικής ευχέρεια των χωρών μελών. Και έτσι δυσκολεύτηκε το σύστημά μας. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι το νέο πακέτο κάνει διαφοροποίηση ανάμεσα στους μηχανισμούς του πυλώνα 2 και την μακροπροληπτική εποπτεία. Είναι πολύ καλό αυτό. Πολλοί όμως παραμένουν σε επίπεδο χωρών μελών που θα ήταν καλύτερο να ασκούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω ότι είναι ένα επίμαχο θέμα. Ε, συζητήσεις γίνονται για τις εξαιρέσεις όσον αφορά τις κεφαλικές απαιτήσει που εφαρμόζονται τώρα σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι ένα από τα εμπόδια στην κυκλοφορία κεφαλαίων μέσα στην Ευρωζώνη. Συχνά λένε τράπεζες ότι αυτό είναι ένα εμπόδιο για αυτή την κυκλοφορία. Ίσως θα έπρεπε όντω να προβληματιστούμε περισσότερο. Είναι κάτι που συζητιέται, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει στις τελευταίες συζητήσεις που έγιναν. Αυτά είναι τα πρώτα που έρχονται στο μυαλό μου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Α, ε, για το θέμα της καταπολέμησης νομοποίησης παράνομων εσόδων δεν είναι στη δικιά μου διεύθυνση, αλλά σίγουρα το να περάσουμε από οδηγία σε κανονισμό θα ήταν μια μεγάλη βελτίωση για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Είναι ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πρόβλημα, οπότε θα έπρεπε να λυθεί και ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλους να ζητούν το λόγο. Οπότε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ νομίζω. Έτσι. Ήταν μια πολύ πλούσια συζήτηση αυτή με πολλά θέματα. Α, στο Catch the Eye έχετε κάτι να ρωτήσετε. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστούμε που είσαστε εδώ υπό τη νέα σας ιδιότητα. Ξέρω ότι την Δευτέρα στους Financial Times δώσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όσον αφορά το τραπεζικό παράγοντα. Και αναρωτιέμαι γιατί ένα από τα πράγματα που είπατε είναι ότι δεν θέλετε καμία πολιτική ανάμειξη και ότι θα φροντίσετε ε, η δουλειά σας να είναι βιώσιμη. Αναρωτιέμαι. Ακούω για δύο τράπεζες που συζητούν για συγχώνευση. και οι οποίε δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχεί σήμερα. Δύο γερμανικέ τράπεζε. Νομίζω καταλαβαίνετε για ποιε μιλάω. Πιστεύετε ότι αν συγχωνευτούν δύο τέτοιε τράπεζε, αυτό θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουν επιτυχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα μεμονωμένα η καθεμία. Τι λέτε γι' αυτό, μπορείτε να παρέμβετε σε αυτό και πώς. Απάντηση. Ναι, δεν ε, βέβαια μπορώ να συμβουλέψω εγώ κυβερνήσεις και δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτό, αλλά αυτό που μπορώ να πω και έτσι απαντάω εν μέρη και σε μια άλλη ερώτηση για τους ε, Ευρωπαίους Εθνικούς Πρωταθλητές. Κοιτάξτε, ο δικός μας ο εποπτικός ρόλος είναι να είμαστε απόλυτα ουδέτεροι, να μην επηρεαζόμαστε δηλαδή από πολιτικά επιχειρήματα. Δεν ε, είμαστε στη θέση μας για να προωθήσουμε εθνικούς ή ευρωπαίους πρωταθλητές. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία πολιτική ατζέντα πίσω από το εποπτικό μας έργο και την αξιολόγησή μας. Ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ούτε καν να συμβουλεύουμε τράπεζα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκτιμούμε ποια είναι τα σχέδια που μας προτείνουν και να τους εξηγούμε ότι από πλευράς ε, εποπτείας ε, θα υπάρξουν αυτά και αυτά τα προβλήματα, κατά πόσο είναι αρκετά ισχυρές για να τα βγάλουν πέρα με ένα τέτοιο σχέδιο, ε, τι θα γίνει με την αποτελεσματικότητά τους, την αποδοτικότητά τους, ώστε να είναι βιώσιμο το σχέδιό τους. Και η ικανότητα επίσης των τραπεζών να έχουν κέρδος και να είναι ελκυστικές επενδυτικά, είναι και αυτό κάτι που παίζει ρόλο εδώ. Αυτά τα στοιχεία είναι που εξετάζουμε εμείς και γι' αυτά ενημερώνουμε και ακριβώς αυτά πρέπει να κοιτούν και οι τράπεζες πριν μας υποβάλουν ένα σχέδιο. Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ να πω. Σβέν εγώ. Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε ιδιωτικό επίπεδο ουσιαστικά γιατί είμαστε πόσοι, τρεις-τέσσερις εδώ. Πολύ ωραία. Θέλω να συνεχίσω μετά από αυτό που είπε η Νίνα Τζιλ. Και θέλω εγώ να το θέσω κάπως διαφορετικά το θέμα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι μία από τις δύο αυτές τράπεζες είναι πραγματικά γερμανική, αν δείτε τη δομή της ιδιοκτησίας, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εντάξει, αυτό το λέω για τους Γερμανούς που ακούνε. Επί της ουσίας όμως και οι δύο τράπεζες για τις οποίες συζητάμε έχουν συγκριτικά και οι δύο εξίσου αδύναμες κεφαλαϊκές θέσεις. Και από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι στην αρχή ακόμα και στις συγχωνεύσεις που ήταν επιτυχής κοστίζει κεφάλαιο μια συγχώνευση. Δεν προσφέρει Μπορεί αργότερα να έρθουν τα κέρδη, αλλά στην αρχή πρέπει να έχεις χρήματα για να μπορέσεις να αντέξεις μια συγχώνευση. Οπότε η ερώτησή μου είναι, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος ως SSM, ως ενιαίος υποπτικός μηχανισμός, σε σχέση με αυτές τις συγχωνευτικές θέσεις. Ξέρετε ότι και ο Γερμανός ο επόπτης στην Deutsche Bank έχει συγκεκριμένη εντολή και είναι αν θέλεις να επηρεάσει τη συζήτηση φώναξε τους, στο, στο κόμμα σου τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Αλλά το γερμανικό κομμάτι της εποπτείας ε, δεν ξέρω κατά πόσο θέλει πραγματικά εντελώ ουδέτερο. Οπότε είναι πιο σημαντικό το τι κάνει ο δικός σας εποπτικό μηχανισμός που είναι ευρωπαϊκός. Οπότε ποιο θα είναι ο δικό σας ρόλος σε αυτή τη διαδικασία ε, συγχώνευσης ή εν πάση συνομιλιών για συγχώνευση. Θα κοιτάξετε την κεφαλική κατάσταση της νέας τράπεζας, γιατί θα πρέπει να απορροφήσει η συγχώνευση ένα μέρο του κεφαλαίου, όπως συμβαίνει συνήθω μετά θα πρέπει να ελέγξετε ποιε θα είναι οι επιπτώσεις στη συνέχεια στην κεφαλαϊκή θέση της νέας τράπεζας. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς το ρόλο σας σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να έχετε ρόλο πολιτικής, αλλά έχετε εποπτικό ρόλο. Και πώς τον ε, εφαρμόζετε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συγχωρείτε, ίσως επαναλαμβάνομαι. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος μας. Δηλαδή κοιτάμε το, το κεφαλιακό, το επιχειρηματικό σχέδιο που μας υποβάλλει η τράπεζα και το εάν έχει κάποιο νόημα και από πλευράς κεφαλαιακής θέσης από το συνδυασμένο κίνδυνο των δύο οντοτήτων εάν τελικά ο οργανισμός ο οποίος θα προκύψει είναι σε μια θέση ώστε να μπορεί μέσω μακροπρόθεσμα να σέβεται τις κεφαλιακές απαιτήσει. Οπότε οπωσδήποτε εστιάζουμε στην κεφαλιακή θέση της τράπεζας. Αυτό κάνουμε σε όλες τις πρόσφατες ε, περιπτώσεις και σε περιπτώσεις στις οποίες οι τράπεζες είχαν ε, δυσκολίες ε, και είχαν κάποια σχέδια, διαρθρωτικά, κεφαλαιακές ενέσεις, προσφορές από άλλες συμμετέχοντες στην αγορά. Ε, αναλύουμε τους αριθμούς και κοιτάμε αν η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι ασφαλής για ένα, σε βάθος χρόνου για να είμαστε όπως είπα σίγουροι για κάτι τέτοιο βεβαίως εξετάζουμε και την κερδοφορία της τράπεζας ε, και το κόστος. Πολλές τράπεζες έχουν ένα κόστος ε, σε σχέση με τα έσοδα πάρα πολύ υψηλό και βεβαίως αυτό επηρεάζει και το πώς εξετάζουμε την συγχώνευση και τους κινδύνους εκτέλεσης της ε, συγχώνευσης. Τη βεβαίως μια πιο περίπλοκη ε, συγχώνευση σημαίνει και υψηλότερου κινδύνου. Και εκεί πέρα θα κάποιε διαβεβαιώσει για το επιχειρηματικό σχέδιο τη τράπεζα. Ναι, παρακαλώ. Ερώτηση. Ανησυχείτε εάν συγχωνευτούν δύο ασθενεί τράπεζε πρώτον και δεύτερον. Ε, είχαν έρθει σε επαφή μαζί σας στα πρώτα στάδια των, ε, της προετοιμασίας. Δεν χρειάζεται να έρθει κανείς σε επαφή μαζί μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις τράπεζες, αλλά ναι βεβαίω, έχουμε ενημερωθεί ότι ξεκινάνε διαπραγματεύσεις, αλλά τώρα περιμένουμε τι διαπραγματεύσεις για να δούμε εάν θα καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια θέση αναμονής βεβαίως ως εποπτική αρχή εμείς πάντα προτιμάμε μια κατάσταση στην οποία έχουμε ισχυρές τράπεζες εξπακούεται αλλά και πάλι δεν θα κρίνουμε εμείς ε, ε, ούτε θα εκφέρουμε κρίση πριν από τις προτάσεις ε, θα πρέπει οι εταιρείε να δουν αν έχει κάποιο επιχειρηματικό νόημα κάποια συμφωνία αν μπορούν να, επιτρέ... να προσελκύσουν επενδυτές. Εμείς την κοιτάμε από την σκοπιά, την προληπτική, την εποπτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μπορεί τώρα να λήξει αυτή η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Ενρία. Επόμενη συνεδρίαση την Πρωταπριλιά στι 3 η ώρα το απόγευμα. Αλήθεια όμως, Πρωταπριλιά αλλά θα γίνει στα αλήθεια.